Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσουμε άμεσα. η είναι κοινά η συνεδρίαση η οποία διεκόπη. Ο κύριος Στίβεν θέλει, κύριος Στίβενσον θέλει να μιλήσει νομίζω για την αντιπροσωπεία στο Ιράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τα νέα σήμερα το πρωί ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ε, απεκάλυψε μία συνωμοσύνη των ε, Ιρανών ε, να δολοφονήσουν το